Ελνοκ. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τα πρακτικά της ε, χτεσινής ε, συνεδρίασης είναι στην διάθεσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά. Εάν όχι, τότε εγκρίνονται. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε τα κατεπήγοντα που αφορούν τις περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Πρώτο ζήτημα είναι η κατάσταση στο Τζιμπουτί. Τον λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ως ένας από τους λίγους βουλευτές που έχει εμπιστευτεί το Τζιμπουτί πρέπει να πω πως έχει πάρα πολλά θετικά. Ε, είναι ένας θαυμάσιος συνδυασμός γαλλικής και σομαλικής κουζίνας και πολιτισμού στην Ερυθρά θάλασσα. Αλλά υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην διακυβέρνηση και η αυταρχική ηγεσία συχνά καταπνίγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες ε, ειδικά των πολιτικών αντιπάλων. Ως εισηγητής για το κέρας της Αφρικής